i submit to you the following changes to the agenda καλημέρα σας ε, κυρίες ε, και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι ε, είχαμε κάποια αναβολή κάποιων σημείων το σημείο 7 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα συζητηθεί στις 10 και 20 το σημείο 8 για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης για την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου Σέγγεν όσον αφορά τη Βουλγαρία και Ρουμανία αναβλήθηκε εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις λοιπόν στην ημερήσια διάταξη όπως αυτή τροποποιήθηκε τότε εγκρίνεται Συνάδελφοι, παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχει διερμηνία σήμερα σε όλες τις γλώσσες ε, και στα ελληνικά. Λιθωνικά μπορείτε μόνο να μιλήσετε, αλλά δεν θα ακούτε. Η συνεδρίαση των ε, συντονιστών ε, μπορείτε να δείτε τα έγγραφα της συνεδρίασης της 20 Μαρτίου στα φάκελό σας. Εγκρίνετε τις συστάσεις των συντονιστών σύμφωνα με το άρθρο 205. Ο χρόνος ψηφοφορίας, η ώρα της ψηφοφορίας έχει οριστεί στις 2 και 5. Στις 10.45 με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ να έχετε μαζί σας την κάρτα ψηφοφορίας. Ξεκινάμε λοιπόν με την κατάσταση στην Ουγγαρία σύμφωνα με το ψήφισμα της 17ης ε, Μαΐου 2017. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 17 Μαΐου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ένα ψήφισμα για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Στην παράγραφο 10 το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή μας να ξεκινήσει την διαδικασία σύνταξη μια ειδική έκθεση για να υπάρξει μια ψηφοφορία στην Ολομέλεια ε, μια αιτιολογημένη πρόταση ε, που καλεί το Συμβούλιο να δράσει συμφώνω προ το άρθρο 7 εδάφιο 1 τη συνθήκη. Ε, σύμφωνα με τον κανονισμό 83 το άρθρο 83 του κανονισμού η κυρία Σαρτζεντίνη ορίστηκε εισηγητής της 11 Ιουλίου 2017 και έκτοτε εργάζεται στην προετοιμασία της έκθεσής της ε, και θα παρουσιάσει σήμερα τα ευρήματά της. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και χαίρομαι πολύ που σας βλέπω να προεδρεύετε σήμερα το πρωί. Συνάδελφοι, ενώ ε, μιλώ, σας μοιράζεται επί χάρτου η έκθεση και ζητώ συγγνώμη για αυτή την ε, ανορθόδοξη αρχή στη συζήτησή μας. Είναι η πρώτη φορά που το Ευρωκοινοβούλιο συντάσσει έκθεση βάσει του άρθρου 7.1. Και για να βεβαιωθούμε ότι όλοι θα λάβουν γνώση, θα φροντίσουμε να μοιραστεί και στους δημοσιογράφους. Και αυτό παρακαλώ σε καμία περίπτωση να μην γίνει πρωτού παρουσιάσω εδώ την έκθεση. Ε, έπρεπε να δείξω κάποια προσοχή στο όλο θέμα, είναι κάπως λεπτό, οπότε καθώς μιλούμε φτάνει στα ηλεκτρονικά σας ταχυδρομεία ε, και mail και θα το δείτε. Είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε και δεν είναι η πλήρης ανταλλαγή απόψεων αυτή, θα ακολουθήσει. Θέλουμε να έχουμε χρόνο, όπως και χρόνο χρειαστήκαμε για να συντάξουμε την έκθεση. Όπως είπατε, Πρόεδρε, αποφασίστηκε το Μάιο του 2017. Έχουμε φτάσει στις 14 Απριλίου. Πολύ καιρό μετά. Είναι μια διαδικασία στην οποία δεν θέλουμε να βιαστούμε. Χρειάζεται χρόνος και προσοχή. Και χρειάζεται και μια διαδικασία ρουτίνας για να γίνεται μια έκθεση αυτή. Κάτι που θα ξεκινήσει τώρα γιατί δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ τέτοια έκθεση. Έχετε λοιπόν μπροστά σας μια έκθεση που βασίστηκε στο παράδειγμα της ε, έναρξη, τη ενεργοποίησης του άρθρου 7 κατά της Πολωνίας. Πρόκειται για ένα ψήφισμα σχετικά σύντομο, αλλά με εκτεταμένο παράρτημα. Θα φτάσω στο περιεχόμενο του παραρτήματος. Επίσης υπάρχει αιτιολογική έκθεση όπου αναλύω τη διαδικασία, τι κάναμε, τι θεωρώ ότι πρέπει να περιλαμβάνουμε τη διαδικασία, ε, σε τι βασίστηκα για να τα προτείνω αυτά που πρότεινα και ότι πρέπει να εργαστούμε προς ε, την επιπλέον σαφήνεια. Ε, εδώ και ένα-δύο χρόνια στο Ευρωκοινοβουλίο αποφασίσαμε ότι ένας εισηγητής ή εισηγητρία μπορεί να συμπεριλάβει υποσημείωση για να ε, εξηγήσει ποιους συνάντησε και με ποιους είχε συνομιλίες και αυτό είναι το τελευταίο τμήμα της έκθεσης. Δεν ε, υπάρχουν αναγκαστικά όλα τα ονόματα στον κατάλογο, αλλά αυτό είναι μια επισκόπηση. Υπάρχουν τέσσερις γνωμοδοτήσεις που θα πρέπει να καλύψει η έκθεση. έχει ψηφιστεί ήδη από την Επιτροπή ΑΦΚΟ. Οι άλλες τρεις έχουν δημοσιευθεί. Της Επιτροπής Ελέγχου των Προπολογισμών, της Επιτροπής Πολιτισμού και τη Επιτροπή ε, για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φίλων. Θέλω να ευχαριστήσω και τι επιτροπέ αυτέ που ανέλαβαν την ευθύνη να συντάξουν και αυτέ ε, την σχετική γνωμοδότηση ε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κάθε μια. Γιατί αυτό ακριβώς θέλαμε να καταλήξει να παρουσιάζει όλη η διαδικασία. Το πεδίο τώρα της έκθεσης και να είμαι τελείως σαφής, διότι είχα πολλές συνομιλίες κατά τη διάρκεια της σύνταξης και κάπως φαίνεται ότι κάποιοι θεωρούν ότι αν ένα θέμα καλύπτεται σε μια διαδικασία με παραβάση η διαδικασία αυτή εφόσον έχει περατωθεί το θέμα αυτό θεωρείται λήξαν. Δεν ισχύει όμως αυτό καθήκον του Κοινοβουλίου και ευθύνη που έχει αναλάβει είναι να εξετάσει πώς όλες οι πτυχές του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί να ε, επιδρούν ε, μεταξύ τους και να σχετίζονται μεταξύ τους. Όπως ε, εξηγώ στο παράρτημα, ακολουθήσαμε τα όσα λέει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου διευκρινίζεται ότι το άρθρο 7 δεν περιορίζεται στο ενωσιακό δίκαιο. Επίσης, εξετάσαμε το τι συμβαίνει στην πράξη. Δηλαδή, ε, είδαμε αν η νομοθεσία έχει ε, αλλάξει, ε, έχει προσαρμοστεί ή έχει επαναχωρήσει, πάντως τα γεγονότα παραμένουν. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε εάν η προτινόμενη νομοθεσία που ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί, έχει οδηγήσει σε μία ε, αποκλιμάκωση της έντασης νομοθεσία που ψηφίζεται, βρίσκεται στο στάδιο της ψήφισή, αλλά ακόμα δεν έχει φέρει τον αντίκτυπό τη στην πράξη. Θα έχουμε μια πλήρη λοιπόν ανταλλαγή απόψεων στη συνέχεια και Εάν καλά θυμάμαι, η υποθεσμένη για την υποβολή τροπολογιών είναι 15 Μαΐου και θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή τον Ιούνιο και στην Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο. Τον Ιούνιο επιδιώκουμε να έχουμε φτάσει σε απλή πλειοψηφία και τον Σεπτέμβριο ελπίζουμε ότι θα έχουμε περισσότεροι. Τώρα, ε, επί των τεχνικών λεπτομεριών, κατέληξα στο συμπέρασμα και μετά από προσεκτική εξέταση όλων των γραπτών εκθέσεων που έχουν συντάξει επιτροπές, ειδικοί απεσταλμένοι, ε, ύπατοι εκπρόσωποι και ενδιαφερόμενοι. Ε, μίλησα μαζί τους και στην Ουγγαρία, στο Στρασβούργο και στη Βουδαπέστη επίση. Και βάσει των όρθρων ορίζει το άρθρο 7 ε, στο πρώτο του εδάφιο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος Παραβίαση των αξιών ε, που αναφέρονται στο άρθρο 2 από ένα κάτω μέλος. Αυτό κοιτάξαμε κατά πόσον μπορεί να ισχύει. Πραγματικά ε, σοκαριστήκαμε όταν είδαμε πόσες προειδοποιήσεις έχουν δοθεί από το 2010 για τόσα πολλά ζητήματα, θα αναφέρω μερικά από αυτά. Είχαμε έξι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις από το 2012 και μετά. Προβλήματα υπήρξαν με το σταματικό δικαστήριο που περιορίστηκε το πεδίο αρμοδιοτήτων του. Τα τακτικά δικαστήρια που ελέγχονται αυστηρότητα, αυστηρότερα από την κυβέρνηση. Έχουν χάσει μέρος της ανεξαρτησίας τους. Η ελευθερία της έκφρασης. Νόμος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νόμος για το παράνομο περιεχόμενο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένα ε, συμβούλιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το οποίο είναι ελεγχόμενο. Ε, ή ε, διαφημίσεις για τους κρατικούς φορείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο ακαδημαϊκός τομέας, η ανεξιθρησκεία, η, από, ε, η αναστολή της άδειας σε εκκλησίες και δόγματα που έχουν εγκριθεί, στα κόμματα, χειραγώγηση της κοινωνίας των πολιτών. Και υπάρχει τώρα και ένας νόμος που πρόκειται να ψηφιστεί και έχει κάποιο αποτελέσματα αποκλιμάκωσης, αλλά υπάρχει και αυτό που λέει ο Ουγγρική Κυβέρνηση Νομοθεσία Όρος. Αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην κοινωνία των πολιτών. Υπάρχει επίσης η υποβάθμιση της ε, όλης ατμόσφαιρας, ε, της ε, ανεκτικότητας που δείχνεται στον πληθυσμό των Ρωμά, τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων επίσης. Πρόεδρε, τα ζητήματα αυτά τα εξετάσαμε ε, επιμέρους και προσεκτικά, αλλά πρέπει να δούμε κατά την αλληλουχία εδώ. Η έκθεση αυτή αφορά το πώς οι Ούγγροι στην Ουγγαρία ε, αντιμετωπίζονται από την ίδια την κυβέρνησή τους. Τα δικαιώματά τους προστατεύονται ακόμα. Έχουν μια κυβέρνηση της οποίας η λειτουργία είναι προβλέψιμη, η οποία έχει κάποια νομική βεβαιότητα στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η χώρα και με τον οποίο συμπεριφέρεται στους πολίτες της. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σοβαρότατη υποβάθμιση των ε, συνθήκων εδώ. Δεν έχει να κάνει με εξωτερικές επιδράσεις αυτό, δεν έχει να κάνει με του δεσάσυλο ή μετανάστες, έχει να κάνει με το δικαίωμα ενός Ούγκρου πολίτη να ε, έχει την μεταχείριση που ο καθένας μας θεωρεί ότι του αξίζει τι θεωρούμε φυσιολογικό. Δηλαδή, θεωρούμε φυσιολογικό το κράτος μου να με προστατεύει. Ε, αυτό είναι το καθήκον που έχουμε ως Ευρωκοινοβούλιο. Να αναλάβουμε δράση και το επισημαίνω και στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δείξουμε ότι οι ευρωπαϊκές αξίες ε, έχουν κάποια σημασία. Κοιτάζω αν έχω κλείσει και ολοκληρώσουμε τις γενικές μου παρατηρήσεις. Πρόεδρε, νομίζω προς στιγμή θα παραμείνω σε αυτά τα σχόλια. Κατανοώ ότι δεν μπορώ να ζητήσω από όλους να το διαβάσουν και να έχουν καταλήξει συνάσματα τώρα αμέσω. Πάντως όλες οι αναφορές που κάνω βασίζονται σε εκθέσεις άλλων. Τίποτε από αυτά που σας ανέφερα δεν είναι προσωπική άποψη της κυρίας Αρχεντίνη. Όλα ε, βασίζονται σε έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει αλλού. Αυτό ε, πραγματικά θέλω να γίνει εδώ είναι να παραμένουμε στα γεγονότα. Και ενώ συνέτασα την έκθεση αυτή, ε, δεν ξεχνάμε ότι είναι πραγματικά, πραγματικά κάτι που μας λυπεί να βλέπουμε ότι πρέπει να βασιστούμε στο Συμβούλιο της Βενετίας, στον ΟΗΕ, σε φορείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φορείς που δεν, μάλλον καθήκοντα που δεν αναλαμβάνουν ε, τα δικά μα θεσμικά όργανα. Στη δήλωσή μου, στην ατυλική έκθεση, υπογραμμίζω ξανά ότι η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το Ευρωκοινοβούλιο να επιζητήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό για το κάτω δικαιώτη, δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι ζωτική σημασία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. ευχαριστούμε για αυτές τις ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις. Να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Η κυρία Μετσόλα, σχεδόν εισηγητής, εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπαμε, η Επιτροπή μας έχει αναλάβει να εξετάσει την κατάσταση στην Ουγγαρία και να παρουσιάσει μια ε, πρόταση και να δούμε κατά πόσον υπάρχει απειλή για την παραβίαση των θεμελιωδών αξιών στην χώρα. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Δεν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε επίθεση κατά τη Ουγγαρία και δεν θέλουμε να ε, γίνει αντιληπτή ω τέτοιο η προσπάθειά μα. Μένουμε στα γεγονότα και θέλουμε να προασπιστούμε το κράτο δικαίου σε οποιοδήποτε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να υπογραμμίσουμε ότι η εκλογική πλειοψηφία δεν δίνει σε καμία ε, κυβέρνηση το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το έχω κάνει και στην περίπτωση τη δική μου πολιτική οικογένεια, ακόμη και αν πρόκειται για την ίδια μου τη χώρα. Και το έχω πει ευθαρσώ. Γι' αυτό λοιπόν, στα πλαίσια αυτή τη συζήτηση, υποστηρίζουμε τι προσπάθειε που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει οι πολιτικές ε, προεκτάσεις να μην ληφθούν υπόψη σε αυτή την προσπάθεια, αλλά να κοιτάξουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες. Θέλουμε να προλάβουμε οποιαδήποτε παραβίαση του κράτους δικαίου με μία προληπτική, με μία ε, προσέγγιση που να βασίζεται στην πρόληψη. Ως προς την έκθεση αυτή, Έχω ασχοληθεί με το θέμα επισταμένος και έχω συμμετάσχει σε όλε τι ε, συνεδριάσεις και οδών και αναεκαθέν υποστήριζα ότι η έκθεση αυτή καλό είναι να είναι συνοπτική και να βασίζεται μόνο σε γεγονότα και σαφείς πληροφορίες. Οποιαδήποτε λοιπόν πολιτική ε, σκέψη ή παραπληροφόρηση δεν έχει καμία ε, θέση σε μια τέτοια έκθεση θεσμικού περιεχομένου. Αναλάβαμε αυτή την αρμοδιότητα με την αντολή που μα έδωσαν οι συναδελφοί μα, αλλά και για λογαριασμό των Ούγγρων πολιτών. Θέλαμε να δούμε την κατάσταση στη χώρα με έναν τρόπο διεξοδικό και χωρί προκαταλήψει. Αυτό ακριβώ έγινε. Όπω σα είπα, θα υπάρξει και άλλη επίσημη παρουσίαση τη έκθεση στην Λίντα, όπου θα έχουμε ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων να εκφράσουμε τις θέσεις μας και τις ιδέες μας με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά η δική μου αρχική αντίδραση είναι ότι υπάρχουν κάποια σημεία που δεν έχουν άμεση σχέση με το κάτω δικαίου στην Ουγγαρία. Βεβαίω, η αδίποτε απειλή στο συνταγματικό σύστημα τη χώρα και ζητήματα όπω η διασφάλιση τη ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου είναι σημαντικά για οποιαδήποτε δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά άλλα σημεία όπω ε, η ε, συμπερίληψη στοιχείων για τα προσωπικά δεδομένα ή η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, κατά την άποψή μα δεν συνάδουν με τον τελικό και τον απότερο στόχο αυτή τη έκθεση. Α μην αναμεικνύουμε διαφορετικά θέματα. Όλα αυτά όμω θα τα λάβουμε υπόψη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι το ε, αποτέλεσμα αυτή τη διαδικασία αντικατοπτρίζει αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην πράξη και να δούμε πώ πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε του πολίτε και να διαφυλάξουμε τι βασικέ αξίε τη Ένωσή μα. Ανυπομονώ για τη συνεργασία μα με την συγκέντρια και του υπόλοιπου συγκητέ. Ε, Ευχαριστώ Ρομπέρτα και τώρα η Άννα Γκόμε, που αντικαστά τον κυρία Βίντιν Χόζερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, χαίρομαι που σας βλέπω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τζουντίθ Σαρτζεντίνη για τη σαφέστατη αυτή έκθεση. Οι εξελίξεις στην Ουγγαρία έχουν οδηγήσει σε ε, σημαντική επιδείνωση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των θεμελιών δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια, όπως ανέφερε ε, με βάση πολλές πηγές μεταξύ των οποίων και εκθέσεις αυτού του Κοινοβουλίου και βεβαίως η ακαδημαϊκή ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον, τον, τον, των μεταναστών, η ελευθερία του συνέρχεστε, ε, η ελευθερία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση, τον, τα δικαιώματα των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες, ε, ε, Εβραίοι, Ρωμά, LGBT, ε, η ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα, η ελευθερία έκφρασης και βεβαίως διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων. Η Όλαφ φέτος υπέβαλε μια έκθεση εξαιρετικά επιβαρυντική ε, για διαφθορά συστηματική ε, προς όφελος της οικογένειας του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και μάλιστα με ευρωπαϊκά κονδύλια. Όλα αυτά ε, είναι μια συστημική απειλή για το κράτος δικαίου. Η δημοκρατία όμως δεν είναι μόνο εκλογές σε ό,τι αφορά τι εκλογέ υπάρχουν άλλωστε σημαντικέ αμφιβολίε για το κατά πόσο οργανώθηκαν δίκαια. Διότι είχαμε απειλέ, είχαμε παρατυπίε σε πάνω από 700 εκλογικά κέντρα. Όλε αυτέ οι παρατυπίε ήταν υπέρ του κόμματο του κυρίου ε, Όρμπαν, την, το Φίντε και της, αποδυνάμωσαν την αντιπολίτευση. Υπήρχε επικάλυψη μεταξύ των πόρων ε, του κυβερνώντος και των κρατικών πόρων κατά τη διάρκεια των της Αυτά λέει η έκθεση της ε, ΟΑΣΕ. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι μετά τις εκλογές από το καθεστώς. Δεν πρόκειται να μετριάσει δηλαδή ε, τη θέση του. Άλλωστε λίγες ώρες μετά ο, ε, ο, ο Ραβίνος ε, της Βουδαπέστης ε, παρετήθηκε. Ένας δημοσιογράφος ε, ε, δολοφονήθηκε, ένας δημοσιογραφικός σταθμός σταμάτησε να εκπέμπει. δεν μπορούμε να σιωπούμε όταν μιλάμε για παραβίαση θεμελιών δικαιωμάτων και αυτών που αναφέρει το αστροδίο της συνθήκης. Η έκθεση τη κυρία Σαρτζετίνη βασίζεται στο ψήσμα τη 17η Μαου, όπου η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου πήρε σαφή θέση κατά τη παραβίαση των αξιών ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε λοιπόν υπέρ τη ενεργοποίηση του άρθρου 7. Εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πάρουμε, παίρνουμε πολύ σοβαρά τις αξίες που αναφέρει το άρθρο 2 τη συνθήκη Συμφωνούμε, υποστηρίζουμε την έκθεση που υπέβαλε η κυρία Σαρτζεντίνη και συμφωνούμε και με την προσέγγιση της. Θεωρούμε ε, ότι βεβαίως υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Δεν, είναι μόνο, δεν υπάρχει μόνο ένας κίνδυνος ε, παραβίασης. Ε, παραβίαση υπάρχει. Υπάρχει συστηματική απειλή ε, για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ήρθε η ώρα το Συμβούλιο να δράσει. Ήρθε η ώρα και η Κομισιόν να δράσει και εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι υπάρχει μόνο μία εξήγηση ε, της αδράνειας αυτής. Ε, το ΕΛΚ προστατεύει τον Βίκτορ Όρμπαν. Μάλιστα, να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Γιούρεκ από την ECR. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαρτζεντίνη. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ε, όταν ήταν και πρόεδρος ε, της Επιτροπής μας ε, και έχουμε βεβαίως εγγύηση της ελευθερίας γνώμης της Τζούντιθ και δικαίως δεν έχω βεβαίω ε, κανέναν λόγο να αμφισβητήσω τις πληροφορίες που μας δίνει. Και ούτε τα συμπεράσματά της. Αλλά όσον αφορά τις ε, πληροφορίες ε, που λάβαμε όταν συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της Ουγγαρίας δεν επιβεβαίωσαν τα λεγόμενα. Εγώ ήμουν σε όλες τις συναντήσεις, έθεσα ερωτήσεις και άκουσα τους ειδικού και τους αντιπροσώπους και ρώτησα αν επιβεβαιώνουν αυτές τις κατηγορίες. Δεν ε, τις επιβεβαιώνουν. Παραδείγματος χάρη η πληροφορία ότι η ΜΚΟ τώρα δυσκολεύονται. Όχι. Μόνο οι ΜΚΟ που λαμβάνουν μεγάλα ποσά από το εξωτερικό πρέπει να ενημερώσουν γι' αυτό. Τι είναι το περίεργο σε αυτό. Θέλουμε να ξέρουμε ποιος, ε, ποιον χρηματοδοτεί στην Ευρώπη ο Πούτιν ή ο Σόρος. Όπως είπαμε ο Σόρος ε, έχει ένα, μια κεντρική δράση η ο σορος οπως ειπαμε ο σορος εχει μια κεντρικη δραση η οποια δεν είναι προβληματική μόνο για την Ουγγαρία αλλά και για το Ισραήλ και για την Ιταλία. Ένα κράτος θέλει να προστατεύσει την κυριαρχία του. Νομίζω ότι μπορεί να ζητήσει αυτές τις πληροφορίες ε, για την χρηματοδότηση. Μετά για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ουγγαρίας. Τι ε, διαπιστώσαμε. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα η παράνομη μετανάστευση. Η Ουγγαρία είχε γνωρίσει τα ίδια προβλήματα με άλλες ε, χώρες. Ένα άλλο πρόβλημα. Η ένταξη των ε, Ρωμά και η εκπαίδευση των, ε, των παιδιών τους. Ε, που είναι ένα πρόβλημα και στα μισά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βεβαίως ε, υπάρχει και πρόβλημα στην Ουγγαρία, αλλά δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Ίσως θα πρέπει να βοηθήσουμε εδώ την Ουγγαρία. Εν ε, Πρέπει να σκεφτούμε αυτό το οποίο είπε η Ρομπέρτα στην αρχή. Η πλειοψηφία δεν έχει πάντα δίκιο και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ούτε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντιλαμβάνομαι ότι αισθάνεται κανείς ε, ευχάριστα όταν ανήκει στην ε, πλειοψηφία. Όπως το λένε οι κοινωνιολόγοι, είναι η αυθεντία που δημιουργείται αν επαναλαμβάνουμε επίσης κάτι συνεχώς ε, τελικά γίνεται αλήθεια. Κατανοητά όλα αυτά, αλλά η πλειοψηφία δεν έχει πάντα δίκιο, ούτε και η πλειοψηφία σε αυτό το κοινοβούλιο. Όσον αφορά τις εκλογές. Πρέπει να εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα. Οι Ούγγροι έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν όπως επιθυμούν υπάρχουν ε, και πολιτισμικές διαφορές. Εμείς ε, θεωρούμε ότι τα δικά μας ε, τα δικαιώματα είναι παγκόσμια και οικουμενικά. Έχουμε άλλες ιστορικές εμπειρίες. Δεν ξέρω μπορούμε να προσδοκούμε το ίδιο από όλες τις χώρες. Σας ευχαριστώ. Κύριος Λουί Η κυρία Ιντεβελτ. Μετά από ο κύριος Γιούρεκ ε, ε, κατά πόσο υπάρχουν πολιτισμικές ε, ή πολιτικές διαφορές μεταξύ πολιτικών κομμάτων, χωρών, ναι βεβαίως. Όμως υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αξιών και μια κοινότητα δικαίου. Και αυτό υπονομεύεται από την κυβέρνηση του κύριου Όρμπαν εδώ και 8 χρόνια. Και θέλω εδώ να υπογραμμίσω, όπως είπαν και άλλοι, ότι εδώ δεν μιλάμε για την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία δεν είναι μόνο ο κ. Σόρμπαν ούτε καν το Φίντες δεν είναι μόνο ο κ. Σόρμπαν Όμως του επετράπει να καταστρέψει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη θεμελιώδη δικαιώματα στη χώρα αυτή. Συμφωνώ με το συμπέρασμα της εισηγήτριας που λέει ότι υπάρχει ένας σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των αξιών πάνω στις οποίες ε, βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πως είναι σαφές για όλους. Ε, δεν είχα την ευκαιρία να διαβάσω το συνόλο της έκθεσης, διότι μόλις, το, μόλις τη λάβαμε, αλλά ε, εδώ μια σειρά από γεγονότα. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, σε άλλα ψηφίσματα. Και κάθε φορά παγιδευόμαστε σε μια κατάσταση, σε μια συζήτηση για το τάδε ή το δίνα μέτρο του κυρίου Όρμπαν που το προτείνει και μετά το αποσύρει. Παίζει ένα παιχνίδι δηλαδή ο κύριος Όρμπαν. Χρησιμοποιεί μια τακτική σαλαμοποίησης, αλλά το αποτέλεσμα τελικά είναι μια συνολική καταστροφή ε, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων. Όπως είπε η ε, είναι αυτή η... Ε, αυτό το αποτέλεσμα που τελικά παγώνει όλους τους τομείς, όλες τις κριτικές ε, φωνές, όλες τις δικλείες ασφαλείας, ε, στον τομέα της εκπαίδευσης ε, αρχίζουν να μαθαίνουν και τα παιδιά να μην έχουν κριτικό πνεύμα, να μην έχουν διαφορετική άποψη έχουν παρθεί μια, σειρά από μέτρα, αλλά υπάρχουν και καμπάνιες μίσους, εκστρατείες μίσους. Ε, ε, είναι πραγματικά ιδιαστικές όταν τις ε, διενεργεί μάλιστα ένας αρχηγός κράτους μέλους της Ένωσης. Μιλάμε για εκστρατείες μίσους. Δεν έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αναρωτηθούμε. Ε, δεν αφορά μόνο το άρθρο 7. εάν η Ουγγαρία αυτή τη στιγμή ήταν υποψήφια χώρα της Ένωσης, θα τη δεχόμασταν. Όχι, δεν θα τη δεχόμασταν. Δεν σοκαριζόμαστε πια όταν η ΟΑΣΕ μετά τις εκλογές ήταν στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν παρατυπίες ε, ε, και ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν δίκαιες οι εκλογές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Θα έπρεπε κανονικά να είμαστε σε κατάσταση σοκ. Και όπως είπε και η Αναγκόμες και η Γιούριθ. Ε, αφορά και τους Ούγγρους πολίτες, τον Ουγγρικό λαό, διότι πέρα από το ηθικό σκέλος ε, του ζητήματος, η διευθυνμένη διαφθορά, η απάτη, το να μην σε γίνουν σεβαστοί οι κανόνες ε, δημοσίων προμηθειών, η κακή χρήση ε, ευρωπαϊκών πόρων και εδώ πρέπει να τα ελέγχει πολύ περισσότερο η Όλαφ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ναι, ναι, τελειώνω. Η κατάσταση αυτή λοιπόν απειλεί την ακαιρεότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη. Ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ και ξέρω βεβαίω ότι το ΕΛΚ είναι διαιρεμένο, ότι υπάρχουν δια... απόψεις διαφορετικές, ότι κάποιοι συνάδελφοι είναι επικριτικοί απέναντι στον κύριο Όρμπαν, όμως το ΕΛΚ προστατεύει τον κύριο Όρμπαν. Ε, τελειώνω ο κύριος Βέμπερ ε, ενθάρρυνε και υποστήριξε τον κύριο Όρμπαν. Και πραγματικά πρέπει τελικά όταν μιλάει για αξίες, να κάνει κάποιες επιλογές. Το άρθρο 7 λοιπόν έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό και ε, υποστηρίζουμε την, ε, την εισηγήτρια. Και τώρα η Μπάρμπαρα Σπινέλη που ε, αντικαστά τη Μαρή στην Βεζιά Ευχαριστώ Παίρνω το λόγο εκ μέρους της κυρίας Βεζιά, η οποία ζητά συγγνώμη από την εισηγήτρια για την απουσία της. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την κυρία Σαρχεντίνη για τη δουλειά της. Ήταν ιδιαίτερα μεθοδική και πάρα πολύ προσεκτική στο να παραμείνει πιστή στα γεγονότα. Έχω εκτιμήσει ιδιαίτερος την επιμέλεια με την οποία συνέταξε την έκθεση ερχόμενοι σε συνεννόηση όχι μόνο με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών αλλά με διεθνείς οργανισμούς που έχουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα ε, στις διάφορες χώρες μας όπως ε, παραδείγματα την Επιτροπή της Βενετίας και την αρμόδια Επιτροπή, τον αρμόδιο φορέα του ΟΗΕ Έγιναν πολλές ακροάσεις και έλεγχοι προς αυτό το σκοπό και πραγματικά ε, η κυρία Βεριζιά ε, εκφράζει την ικανοποίησή της για αυτό. Οι έλεγχοι αυτοί έδειξαν ε, ξεκάθαρα ότι το επίπεδο ανησυχιών των πλέον σημαντικών διεθνών οργανισμών είναι δικαιολογημένο. Η δική τους αποτίμηση θα μπορούσε συνοπτικά να δοθεί ως εξής από καιρό το κράτος του δικαίου κινδυνεύει και απελείται στην Ουγγαρία και πλέον μπορεί να χαρακτηριστεί συστηματική και μόνιμη αυτή η απειλή. Και προ στιγμή τα πράγματα δεν βελτιώνονται. Ο τελευταίος νόμος για τις μη κυβερνητικέ οργανώσει που ασχολούνται με την ένταξη των ε, μεταναστών, που παρουσιάστηκε στι ε, αμέσω πριν τι εκλογέ, είναι κατά την άποψη των οργανισμών αυτών επικίνδυνος διότι προετοιμάζει και ε, μάλλον θέτει να αμφιβόλο όλη αυτή τη δουλειά ε, υπέρ της ένταξης που είναι και προς όφελος της Ουγγαρίας και της κοινωνικής της συνοχής. Τα αποτελέσματα των εκλογών ξέρουμε από την ιστορία μπορούν ε, να είναι έτσι ή αλλιώς όμως παραμένει ερώτηση, απορία κατά πόσον υπάρχει παραβίαση του κράτους δικαίου ή όχι. Και η απορία αυτή πρέπει να απαντηθεί. Ακόμη και αν είναι ευνοϊκό το αποτέλεσμα των εκλογών υπέρ αυτού που παραβίασε το κράτο δικαίου. Ένα άλλο σημείο που θέλει να υπογραμμίσει η Μαρή Κριστίν Βερζιά είναι το εξή. Από το 2010 το Ευρωκοινοβούλιο απευθύνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση για την προάσπιση του κράτου δικαίου στην Ουγγαρία. Η ε, διστακτικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτά τα 8 χρόνια δεν εξυπηρέτησαν τον σκόπο μας, διότι ουσιαστικά υποδάβλησαν ε, την καχυποψία προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Και υπήρξε παρεκτροπή ως προς το κάτω δικαίου και σε αυτές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγώντας σε μια γενικευμένη υποβάθμιση στην ε, Ένωση. Και είναι πραγματικά ε, δηλητηριώδεις αυτές οι στρατηγικές, μπορεί να έχουν δηλαδή αποτέλεσμα ε, μοιραίο, ε, ως προς το πώς αντιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οι πολίτες των χωρών αυτών με τη δράση των ε, κυβερνώντων της χώρας αυτές. Είναι κάτι που δεν πρέπει να συμβεί. Η ε, αποτίμησή μα για τα διάφορα κράτη-μέλη όμω πρέπει πάντοτε να είναι αντικειμενική και αμερόληπτη, όποιε και αν είναι οι συνθήκε. Η ορολογία ε, και η μέθοδο που ακολούθησε η Γιούντιτ Αρχεντίνη είναι εξαιρετική. Γι' αυτό θα μελετήσουμε την έκθεση. Η Μαρή Κριστίν θα διαβάσει προσεκτικότατα την έκθεση και θα δει αν είναι σε θέση να υποβάλει τροπολογίε. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα κύριος ε, Λεμπρετών που αντικαθιστά τον κύριο Μπάι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση αρχεντίνη είναι σημαντική διότι ε, λαμβάνει ε, ως αφετηρία την ενεργοποίηση του άρθρου 7 κατά της Ουγγαρίας. Κάτι μπορεί να ε, στερήσει τη χώρα αυτή από κάποιες από, τις, ε, από τα Θα ήθελα να δώσω τρία ε, παραδείγματα εδώ για τις επικρίσεις κατά της Ουγγαρίας. Εδώ ε, καταδικάζουμε την Ουγγαρία για τον νόμο κατά του Σόρος, όπως ονομάστηκε, Stop Σόρος. Δεν είναι όμως λογικό ένα κράτος να θέλει να ελέγξει τη χρηματοδότηση κάποιων οργανώσεων που μπορεί να έχουν και ρόλο ε, ακτιβιστών ε, στην επικρατεία της. Εδώ αμέσως υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει ανάμειξη της Ρωσίας και αμέσως ανεβάζουμε τους τόνους, όμως στο στόχαστρο βρίσκεται ο Σόρος και τότε βρίσκουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να λάβουμε δράση. Εγώ υποστηρίζω την Ουγγαρία στην πρόθεσή της, στη βούλησή της όπως την έχει εκφράσει ευθαρσός, να ε, υπερασπίσει τον εαυτό της σε σχέση με όσα γίνονται στην επικρατεία της. Δεύτερο παράδειγμα, η Ουγγαρία έχει ε, υψώσει ε, νέα τύχη και ουσιαστικά σκέφτεται το έλεγχο στα σύνορά της με τη Σλοβακία και την ε, Σερβία. Από το 2015, 140.000 μετανάστες, ε, παράνομοι μετανάστες, έφτασαν σε ένα μήνα την, στην Ουγγαρία. Τι περιμένετε από μια χώρα που δεν έχει τεράστιο πληθυσμό ε, όπως η Ουγγαρία. Είναι ε, απόλυτα λογικό να έχει ξεκινήσει αυτό το φράξιμο των συνόρων ε, για να προστατευτεί. Κάθε κράτος έχει δικαίωμα να προστατεύσει την ταυτότητά του. Εδώ λοιπόν και πάλι συμφωνώ με όσα κάνει η Ουγγαρία. Τώρα το φαινόμενο της μετανάστευσης ξεπερνά την ίδια την Ουγγαρία και αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε ε, από κοινού και όχι μόνο να κατηγορήσουμε και να απομονώσουμε την Ουγγαρία. Επίσης το σχέδιο επανεγκατάστασης των μεταναστών, το περίφημο σχέδιο Κέρο που δεν θέλει να συμμετάσχει η Ουγγαρία. Τρίτο παράδειγμα, εδώ δεν μπορούμε να τις ε, ε καταλογίσουμε κάτι, διότι είναι απόφαση του Ουγγρικού λαού. Δημοψήφισμα έγινε και τα συντριπτική πλειοψηφία του λαού τοποθετήθηκε κατά του προγράμματος αυτού. Επίσης ο κύριος Ορμπάν κέρδισε θριαμβευτικά τις ε, βουλευτικές εκλογές. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε εφόσον ο λαός εκφράστηκε. Πρέπει να σεβαστούμε την δική τους κυρίαρχη βούληση και επιθυμία. Ε, σας ευχαριστώ. Η κυρία Φερέρα ενθουσιάζει. Η κυρία Βίνμπερκ λοιπόν θέλει το λόγο από το EFTD. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Σαρτζεντίνη για την έκθεση αυτή. Ε, παρά το ότι μας την έστειλε κάπως αργά και δεν προλάβα να τη διαβάσω ολόκληρη. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί εδώ μέσα ανησυχείτε για το ότι η Ουγγαρία δείχνει τον δρόμο για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους Ούγγρους για τα αποτελέσματα των εκλογών, την στήριξη στον Βίκτορ Όρμπαν και αντιλαμβάνομαι ότι ενισχύεται βεβαίως. Ο κόσμος ε, είναι ενθουσιασμένος, υπερασπίζεται τους ε, νέους, ε, υπερασπίζεται τα σύνορα της χώρας του, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι ανησυχείται κάπως με αυτές τις εξελίξεις. Αντιλαμβάνομαι ότι η Ουγγαρία αντιμετωπίζει κάποιε προκλήσεις, όλες οι χώρες όμως, όλα τα κράτη-μέλη. Η Ρωμά, η ένταξη των μεταναστών, τέτοια θέματα υπάρχουν σε πολλές χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ειδικά στο θέμα της ένταξη των μεταναστών. Δείτε τις χώρες που δέχτηκαν τεράστιου αριθμού. Η Ουγγαρία λέει ότι αν δεν μπορούμε να τους ε, εντάξουμε δεν θα πρέπει να δεχτούμε τόσους πολλούς. Ε, νομίζω πρέπει να τους σεβαστούμε αυτό και να συγχαρούμε την Ουγγαρία για τις ε, δημοκρατικές εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην Κίνγκα Γκάλε. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Θα προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω πως είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής από το 2004 και από το 2007 αντιπρόεδρος, αλλά βλέπουμε ότι τέτοιες διαδικασίες δεν είχαμε ποτέ. Ποτέ δεν έχουμε συζητήσει μια τέτοια έκθεση ε, και να την λαμβάνουμε λίγο πριν την ε, έναρξη της συνεδρίασης. Κανείς δεν έχει μπορέσει να διαβάσει ε, εις βάθος την έκθεση της Αργεντινή, αλλά πρέπει να σας πω ότι η εφημερίδα Νύψοβο είχε διαβάσει το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης παρά το ότι η κυρία Σαρτζεντίνη ε, είπε ότι δεν θα είχε συντάξει την έκθεση πριν τις εκλογές και όμως είχε διαρρεύσει η έκθεση. αν είχαμε λίγο χρόνο αλλά την διάβασα. Λοιπόν, ε, άκουσα προσεκτικά την συζήτηση και θα ήθελα να τονίσω πως η βάση του κράτους δικαίου είναι το αποτέλεσμα των δημοκρατικών εκλογών. Όσο δεν δεχόμαστε το αποτέλεσμα των εκλογών δεν μπορούμε να μιλάμε για κράτος δικαίου ανεξαρτήτως του τι λέει η κυρία Ινετφέλτ. Ο ΟΑΣΕ δεν αμφισβήτησε την εγκυρότητα των εκλογών. Ο τύπος, η τιμένη αντιπολίτευση ε, θα ήθελε να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Να επαναλάβω λοιπόν η Ουγγαρία δεν πρέπει να προστατευτεί όπως λέτε παρά τη θέλησή της. 70% των πολιτών ψήφισε και ε, έδωσαν το αποτέλεσμα. Δηλαδή αν δεν είναι αυτό δημοκρατία τι είναι. Αν δεν σας αρέσει η δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία πια και δεν είναι κράτος δικαίου αυτά είναι υποκειμενικά συναισθήματά σας. Γιατί θέλετε ε, μια συγκεκριμένη πολιτική και να δεχτούμε υποχρεωτικά μετανάστες. Αυτό είναι εκστρατεία μίσους, αυτό το οποίο διεξάγεται κατά της Ουγγαρίας. Στην ε, Ουγγαρία δεν χτυπάει η αστυνομία ε, διαδηλωτές ε, δεν ε, συλλαμβάνει δημοσιογράφους και όμως μόνο στην Ουγγαρία βλέπετε εσείς τέτοια προβλήματα. Πώς είναι δυνατόν όλα τα προβλήματα να υπάρχουν μόνο στην Ουγγαρία. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία έχουν απαντηθεί επαρκώς ή έχουν επιληθεί θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω. Ε, πραγματικά αισθάνεστε ότι ξέρετε καλύτερα την κατάσταση στη χώρα από τους ψηφοφόρους που ζουν εκεί. Ναι, ναι, τελειώνω. Εάν λοιπόν μπούμε λίγο πιο βαθιά σε αυτήν την έκθεση, βλέπουμε συνεχώς τις ίδιες ΜΚΟ, συνεχώς τα ίδια δημοσιεύματα. Πρόκειται δηλαδή για μια δίκη παροδία όπου έχει ληφθεί η απόφαση, η πολιτική απόφαση από πριν και δεν λαμβάνουμε υπόψη τα γεγονότα. Ε, Κύριο Σέγγελ για δύο λεπτά. Θα προσπαθήσω. Δεν είναι το πρώτο έγγραφο που αφορά την Ουγγαρία αυτό που έχουμε μπροστά μπροστά μας. Ε, ε, πολλές φορές στο παρελθόν ε, έχει γίνει το ίδιο λάθος. Επικεντρωνόμαστε πολύ στα αποτελέσματα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν ο Ραβίνος παρετήθηκε. Διότι δεν νομίζω αυτό να έχει να κάνει με το πρόβλημα του αντιστημιτισμού στην Ουγγαρία. δεν με νοιάζει πόσες είναι οι αναγνωρισμένες εκκλησίες στην Ουγγαρία. Είναι πάντως περισσότερες από ό,τι στο Λουξεμβούργο. Αλλά δημιουργείται εδώ μια ατμόσφαιρα ε, η οποία οδηγεί στο να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Ουγγαρία, στις εκλογές. Η μισή από τους εκλογείς, από τους ψηφοφόρους που προσήλθαν στις κάλπες, ψήφισαν ε, φίντες. Άλλο 20% ψήφισε Ιόμπικ. Μένει ένα 30% που ψήφισε ε, μια αντιπολίτευση όχι τόσο αξιόπιστη, πράσινοι σοσιαλιστές. Ε. αυτό είναι το το πολιτικό τοπίο, ε, αυτό το οποίο διαμόρφωσαν, διαμόρφωσαν οι ψηφοφόροι. Υπάρχει όμως λόγος γι' αυτό. Έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα τα τελευταία χρόνια. Ε, το κλίμα ότι άλλαξε το κράτος. Όταν ήρθε το 2010, όταν ήρθε το 2010 ε, στην εξουσία ο, Όρμπαν, ε, είπε ότι δεν θα κάνει τα λάθη που έκανε το 1998 και το 2002 όταν έχασε τις εκλογές, όταν τον κέρδισαν, είπε ότι πρόκειται να ξανακάνει ε, το ίδιο λάθος, δεν θα υπάρχει κανείς αρκετά ισχυρός απέναντί του για να τον κερδίσει. Και έγιναν, χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα, η κάθε προσπάθεια για να μην βρει αντίπαλο ξανά στο πολιτικό σκηνικό. Είναι λίγο δύσκολο αυτό βέβαια ε, να συμπεριληφθεί σε μια έκθεση άρθρο 7. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Είναι ένα κλίμα εντός του οποίου κάποιος που θέλει να δώσει την ευκαιρία σε νόμιμους μετανάστες να εργαστούν ε, του σκιάνε τα λάστιχα και τον απειλούν οι συγχωριανοί του απλώς ε, βρέθηκε εντός της κατηγορίας ε, ανθρώπων που ε, στοχοθετεί, στοχοποιεί η προπαγάνδα του Φίντες. Εγώ δεν θα ήθελα να στείλω κανένα μετανάστη στην Ουγγαρία. Διότι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν. Όχι λόγω της Εκκλησίας, αλλά επειδή το κόμμα που κυβερνάει αυτή τη στιγμή στην Ουγγαρία αποφάσισε κάποια στιγμή ότι ε, η ύμνη ε, στην Ουγγρική ταυτότητα είναι το μόνο πολιτικό πρόγραμμα. Και το κράτος πλέον βασίζεται στο μίσος. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα κράτος να, να, να στηρίζεται στο μίσος. Και πρέπει να μπορέσουμε αυτό να το συμπεριλάβουμε στην τελική εκδοχή της έκθεσης της Γιούριθ. Είναι λίγο δύσκολο από νομικής πλευράς βέβαια, αλλά αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ο αριθμό των αναγνωρισμένων εκκλησιών, δεν είναι ο κύριο όρο, δεν είναι η κεντροευρωπαϊκή, το κεντροευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, δεν είναι αυτά τα ζητήματα. Ακόμα και αυτά που περιλαμβάνουν στη διαδικασία σε παραβάση. Είναι η δημιουργία μια συνείδηση ενό κλίματο, μάλλον η συνειδητή δημιουργία ενό κλίματο, ε, όπου διώκεται οτιδήποτε δεν χωράει, δεν ταιριάζει σε αυτό το αφήγημα. Και αυτό δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπιόρκη ένα λεπτό παρακαλώ, διότι πρέπει να ψηφίσουμε. Θα είμαι σύντομη. Ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της και ότι βασίστηκε στις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες, στις ε, δημοκρατικές αρχές ε, και συμφωνώ και με αυτό που είπε ο τελευταίος ομιλητής. Είναι σημαντικό. Έτσι πρέπει να εργαστούμε να δούμε τις λεπτομέρειες όμως, να δούμε τις λεπτομέρειες ε, ε, των δράσεων, των πράξεων μιας τέτοιας κυβέρνησης ε, και οι επιπτώσεις για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Και εμείς εργαζόμαστε επί αυτής της έκθεσης στην Επιτροπή Γυναικών. Η κυρία Νόσπερκ είναι η συγκήτρια και θα συνεισφέρουμε και εμείς, διότι η κατάσταση και για τα για τους υπερασπιστές των, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών ε, στην ε, Ουγγαρία είναι δύσκολη. κυρία Γιώκα, ευχαριστώ πολύ. Να κάνω και εγώ, λέει κυρία Γιαρόκα, κάποια σχόλια. Καταρχήν είναι σκανδαλώδες ότι προσπαθούμε εδώ ε, να χρησιμοποιήσουμε τους Ρωμά για να πλήξουμε την Ουγγρική κυβέρνηση. Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι αυτός που έστειλε τον πρώτο Ρωμά Ευρωβουλευτή ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι αυτή και χάρη στον Ουγγρικό λαό είμαι εδώ σήμερα. Χάρη στους συναδέλφους μου, χάρη στην Ουγγρική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Ρωμά μπόρεσε να προχωρήσει στις Βρυξέλλες. Θετικά παραδείγματα υπάρχουν πολλά χωρίς την Ουγγρική κυβέρνηση δεν το είχαμε πετύχει αυτό. Η εβδομάδα των Ρωμά που οργανώθηκε στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα με τους εμπειρογνώμονες ε, που προσκλήθηκαν. Δεν θα μπορούσαν να γίνει αυτή η εβδομάδα, αυτή η εκδήλωση χωρίς όλες αυτές τις επιδοτήσεις, τις ενισχύσεις, εάν η Ουγγρική κυβέρνηση και άλλα κρατημέλη δεν είχαν ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία. Αν οι συνάδελφοι σοσιαλιστές ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το θέμα, οπότε δεν θα είχαν ψηφίσει, δεν ψηφίσει κατά της πρότασής μας ε, να εξεταστεί για άλλη μια φορά το θέμα αυτό. Και απλά να έχουμε μια ακρόαση όπου καθένα διαβάζει τις ομιλίες του. Λοιπόν, κυρία Συγήτρια, η έκθεσή σας ε, περιλαμβάνει ψευδή στοιχεία. Λέτε ότι γίνονται, ε, ε γίνονται παρελάσεις της ε, Ουγγρικής φρουράς ε, ενώ ε, έχουν απογορευτεί από τον κύριο Όρμπαν ενώ επί σοσιαλιστικής κυβέρνησης έχουν δολοφονηθεί Ρωμά τότε ναι, τότε φοβόντουσαν ε, ε, οι Ρωμά όταν έκαναν αυτά τις παρελάσεις στις Ουγγρικές φρουρές και οι Ρωμά κατά πλειοψηφία ψήφισαν φίντες είναι το Φίντες που επέτρεψε στις, στους, στους Ρωμά να έχουν πρόσβαση σε μια σε μια αξιοπρεπή στέγαση. 220.000 άνθρωποι βρήκαν θέσει εργασία υπό τον Όρμπαν. Μπορούσαν να βρουν κατάρτιση. Και μέσα και έχω το λόγο να σα πω και το εξή. Εάν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τόσο σημαντικά για τα θεσμικά μας όργανα, θα πρέπει να ακούσουμε και τον κύριο Λεγκλόντ. όχι να τον διώξουμε μετά από μία μέρα επειδή, ε, επειδή κριτήκαν τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ για ένα λεπτό. Ένα λεπτό νομίζω ότι είναι διακριτική μεταχείριση εις βάρος μου, αλλά τέλος πάντων. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Έγγελ, ο οποίος πολύ καλά συνόψε την κατάσταση. Περί τίνος πρόκειται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί ε, την Ουγγαρία ως άκου του box, διότι έχουμε παρουσιαστεί ως κακοί μαθητές. Δεν ε, θέλουμε μετανάστες, δεν θέλουμε ποσόστοση, δεν θέλουμε μαζική μετανάστευση στη χώρα μας. Και κατά την άποψή μου δίνουμε ένα παράδειγμα όλοι τα κράτη-μέλη. Τους δείχνουμε ότι υπάρχει και άλλη εναλλακτική λύση, ότι μπορούν οι λαοί τη Ευρώπη να διατηρήσουν ε, την ελευθερία τους, γιατί και εμείς χρειάστηκε στην αρχή να αντιμετωπίσουμε τεράστιες ε, αντιστάσεις. Πάμε και με ανάντια στο ρεύμα και προσπαθούμε να αντισταθούμε σε αυτά που προσπαθεί να μας μεγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας θυμίζω ότι 75% του πληθυσμού στήριξε την κυβέρνηση Όρμπαν στο πρόσφατο δημοψήφισμα για τη μεταναστευτική του πολιτική. Θα ήθελα πάντως εδώ να σας ευχαριστήσω κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω την ε, κυρία Ιντφελτ, η οποία δεν ξέρει καθόλου τι γίνεται στι σχολέ νομική τη Ουγγαρία, αλλά μιλάει λε και είναι ειδική επί του θέματο και έχει αποφετήσει από νομική σχολή στη χώρα μα, και την κυρία Σαρχεντίνη, που κρίνεται την ε, ε, χώρα μα και απευθύνεστε στην Ουγγαρία, κάνοντά την μια χώρα δακτυλοδεικτούμενη με ένα σωρό κατηγορίε. Εδώ στην ε, ε, αίθουσα έχουμε ένα σωρό βουλευτές και βοηθούς και άλλο πολύ κόσμο, αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν νοιάζεται εδώ στην αίθουσα. Οι συνάδελφοι φαίνεται να μην έχουν κάνει καν τον κόπο να έρθουν σε αυτή τη συνεδρία γιατί βαριούνται απλώς. Ε, θέλετε την πλατεία Μαϊντάν και τις διαδηλώσεις της, θέλετε την Αραβική Άνοιξη, αλλά στην ουσία ε, έχουμε εδώ μια Ε, η Ουγγαρία μπορεί να γίνει μια δεύτερη Μαϊντάν αν επιμείνεται, αλλά δεν το θέλουμε αυτό. Να κοιτάξουμε να επιδιώξουμε τη σταθερότητα και την ε, ηρεμία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι αναπληρωτής ε, εδώ. Δεν σκόπευα να πάρω το λόγο, αλλά θέλω να επιμείνω, γιατί και εγώ είμαι πατέρας ε, οικογένειας, είμαι πατριώτης και είμαι υπερήφανος. Πραγματικά ντρέπομαι. Ε, ντρέπομαι σήμερα, διότι η Ουγγαρία έχει φτάσει σε αυτήν την θέση λόγω των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία λεπτά είδατε λιγάκι τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι της Φίντες και βλέπετε τα ψεύδη που ακούγονται κατά της χώρας. Η Ουγγρική κοινωνία για άλλη μια φορά ε, είναι αυτή που έχει πέσει στην παγίδα διότι ε, ο κύριος Όρμπαν και οι φίλοι του έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν όπως θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε τι γίνεται εδώ κυρίες και κύριοι. Το Φίντες κατά την έκθεση της κυρίας Σαρχεντίνη και όσων ε, ε, ακούστηκαν σήμερα εδώ, εκδικείται την Ευρωπαϊκή Ένωση με το αποτέλεσμα των εκλογών την Κυριακή. Εμείς όμως φροντίσαμε η έκθεση αυτή να συζητηθεί αμέσως μετά από τις εκλογές της Κυριακής για να μην θεωρηθεί ότι υπάρχει κάποια επίδραση στο εκλογικό σώμα. Ε, πραγματικά ντρέπομαι για όσα ακούγονται πάντως εδώ σήμερα. Ε, λόγω των εσωτερικών ε, πολιτικών πραγμάτων στη χώρα μου, την Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Να σας ενημερώσω ότι η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης θα γίνει στις 25 και 26 Απριλίου όταν θα ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις. Ε, κύριε Σαρτζεντίνη, θέλετε να συνοψίσετε. Σας ευχαριστώ. Όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσω να συνοψίσω την συζήτηση. Βεβαίω, ε, χαίρομαι όταν συνάδελφοι θέλουν να βελτιώσουν την έκθεση. Θα συνεχίσει η διαδικασία να είναι διαφανής. Και χαίρομαι που οι συνάδελφοι αναγνωρίζουν το πώς ε, εργαστήκαμε. Αλλά δεν έχει νόημα να αρχίσω να σχολιάζω τις απόψεις των ε, συναδέλφων. Έχουμε γνώμη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Θα περιμένουμε λοιπόν ε, την 25η Απριλίου. Περνάμε στο σημείο 4. Ερώτηση προς την Κομισιόν ε, της 24ης Οκτωβρίου 2017 από την Σόφη Ινετφέλτ για την έλλειψη ανεξαρτησίας ε, της πολωνικής δικαιοσύνης και το πώς θα επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία. Συνάδελφοι, περνάμε σημείο 4. Η κυρία Ινετφέλτ είναι η συντάκτης. Και σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 5 του κανονισμού η προθεσμία για γραπτή απάντηση είναι 6 εβδομάδες. Λάβαμε την απάντηση της ε, Κομισιόν μόλις στις 7 Μαρτίου 2018. Οπότε, σύμφωνα με το άρθρο 5, με το εδάφιο 5 του άρθρου 130 του κανονισμού, οι συντονιστές της ΛΥΜΠΕ αποφάσισαν να, ε, να μπει το θέμα αυτό στη μέση διάταξη της Επιτροπής μας. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην συντάκτη. Η κυρία Ίνετφελντ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι η Κομισιόν μου έστειλε ε, μια απάντηση. Σε Μαρτίου. στην ουσία δεν πρόκειται περί απάντησης. Όπως ε, συνήθως συμβαίνει με την Κομισιόν, η ουσία της ερώτησής μου είναι η εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεράνει ότι η έγκριση διαφόρων νόμων από το Πολωνικό Κοινοβούλιο αυξάνει την συστημική απειλή στο κράτος δικαίου, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτό θα επηρεάσει την αστυνομική ε, συνεργα... και δικαστική συνεργασία. Παραδείγματο χάρη, όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη, ένταλμα έρευνα, αλλά και την αξιοπιστία των δεδομένων που θα βάζει στις διάφορες βάσεις δεδομένων η Πολωνία, όπως το ΣΥΣ ε, κτλ. Και καθώς πηγαίνουμε προς την ίδια λειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα, από την επόμενη εβδομάδα θα μιλάμε για ηλεκτρονικά στοιχεία στις δίκες θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι δικαστικές αρχές είναι πλήρως ανεξάρτητες. Τώρα, πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι όλα αυτά είναι κάποια αριστερή συνωμοσία. Τώρα όμως ένας Ιρλανδός δικαστής απέρριψε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ε, των Πολωνικών Αρχών λέγοντας ότι στην Πολωνία, λέει ο δικαστής, έχει υπονομευθεί συστηματικά το κράτος δικαίου και παραβιαστεί η δημοκρατία. Το Ιρλανδικό Δικαστήριο παρέπεμψε το ζήτημα στο ΔΕΚ. Οπότε ήδη έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα πλέον. Είχαμε τη συζήτηση με την Ουγγαρία, τώρα μιλάμε για την Πολωνία. Τα πράγματα γίνονται πραγματικότητα. Και θα επεκταθούν, είμαι σίγουρη. Η περίπτωση αυτή λοιπόν αποδεικνύει γιατί είναι σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη να πληρούν κάποιες προδιαγραφές ε, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να λάβω μία απάντηση εγώ από την Κομισιόν και βεβαίως θα λάβουμε μια, απόφαση, μια απάντηση από το δικαστήριο τώρα, αλλά αυτό το οποίο έχει πει η Κομισιόν είναι ότι έχουμε μια διαδικασία του άρθρου 7. Αυτό δεν είναι απάντηση. Η Κομισιόν είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και αυτό ε, έχει κάποιες επιπτώσεις εδώ πέρα βλέπετε στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και Έρευνας. Θέλω να μάθω από την Κομισιόν ποιες είναι αυτές οι συνέπειες. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιο άλλο τον λόγο. Η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στην Σόφη που πρόβλεψε να τεθεί η ερώτηση αυτή και είμαι και εγώ ιδιαίτερα απογοητευμένη με την απάντηση που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι λέει η Επιτροπή ότι ενδιαφέρεται ίσως να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του άρθρου 7, διαδικασία επί παραβάση. Ωραία. Όμως το εμπροκειμένο ερώτημα που θέτει η Σόφη Ιντβέλτ δεν έχει απαντηθεί και ούτε εγώ ε, βρίσκω απάντηση σε αυτά που λέει η Επιτροπή. Τι νόημα έχει να έχουμε τόσα θεσμικά όργανα, τόσους οργανισμούς που ασχολούνται με την οικονομική συνεργασία και την καλλιεργούν και να δημιουργήσουμε και θέλουμε να δημιουργήσουμε και νέους φορείς εάν δεν μιλάμε για χώρες όπου το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών δεν τηρούνται 100%. Τι νόημα έχει να επιδιώκουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον Ευρωπαίο Εισαγγελία, εάν δεν γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου και ο διαχωρισμός των εξουσιών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ λοιπόν και στηρίζω τη μάχη της Όφη για το θέμα αυτό και πραγματικά αναμένω διακαώς μία ε, πραγματικά διεξοδική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. πάλι στο εδόλιο η εθνική κυριαρχία και οι χώρες ε, που ε, θέλουν να βάλουν στη θέση του κατηγορουμένου την Ουγγαρία, τη χώρα μου, όπως ακούσαμε νωρίτερα σήμερα και δεν μας εκπλήσει αυτό βεβαίω και την Πολωνία. Ήθελα εδώ να επιστήσω την προσοχή των ε, Πολωνών φίλων. Έχουμε αυτή τη στιγμή 8 ευρωβουλευτές στην αίθουσα. Και ετοιμαζόμαστε να λάβουμε ενδεχομένω αποφάσει που ίσως να καταλήξουν ε, στο πέρα της διαδικασία σε σοβαρέ κυρώσει. Έχουμε εδώ επισκέπτε, συνεργάτες μας από τη διοίκηση, βοηθούς, ε, εκπροσώπους άλλων θεσμικών οργάνων και από του εκατοντάδε βουλευτέ του θεσμικού αυτού οργάνου, πόσοι ευρωβουλευτέ ενδιαφέρονται για την έκθεση αυτή, οκτώ. Να είμαστε σαφεί. Ό,τι η Πολωνία, ό,τι η Ουγγαρία θα έπρεπε να έχουν ε, ε, πέσει στα χέρια αυτή τη μικρή ομάδα για να κρυθούν. Έχουμε τον πολιτισμό μας, την οικονομία μας, ε, την κυριαρχία μας και είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας. Δεν μπορείτε να μας κοροϊδεύετε διαρκώς. Δεν μπορείτε να παίζετε με μια χώρα όπως ε, η Πολωνία ούτε με την Ουγγαρία και να σας διαβεβαιώσω ότι στη δική μας, στις δικές μας χώρες υπάρχει εθνική ενότητα και υπάρχει και αντίσταση η οποία διαρκώς ενισχύεται ε, λόγω των επανειλημμένων προσπάθειών σας να μας ταπεινώσετε. Και για την Ουγγαρία και για την Πολωνία ισχύει αυτό. Πρόεδρος, επειδή με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ε, κυρία Μορβάη, επειδή δεν είστε τακτικό μέλος αυτής της Επιτροπής, δεν είστε καν αναπηρώτρια να σας επισημάνω ότι η ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και τους δικηγόρους έγινε πριν από μια μισή εβδομάδα περίπου συζητήθηκε με τη συμμετοχή πολλών ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο εφόσον θέλει. Please, colleagues. Please, colleagues. Σας παρακαλώ τη συνάδελφοι, η κυρία Ρίγκου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να σας δώσουμε κάποια περαιτέρω στοιχεία για ε, το κοινοβουλευτικό ερώτημα της αξιότιμης ε, κυρίας Σίντεβελ, Βέβαια θα λάβει την απάντησή μας και γραπτός. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι η ανεξαρτησία των κρατών μελών και των δικαστικών συστημάτων είναι κρίσιμη σημασία για την αμοιβαία εμπιστοσύνη σε ζητήματα δικαιοσύνη και ιστορικών υποθέσεων. Είναι επίση κρίσιμη σημασία για την ορθή εφαρμογή των νομοθετικών μέσων της Ένωσης που βασίζονται σε αυτή την εμπιστοσύνη. Η έλλειψη εμπιστοσύνης του δικαστικού τομέα σε ένα κράτος μέλος, η έλλειψη μάλλον ανεξαρτησίας, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' τον το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να αντιμετωπίσει την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Η σημασία του κράτους δικαίου για την αμοιβαία εμπιστοσύνη στον τομέα δικαιοσύνης και αστυνομικών υποθέσεων υπογραμμίστηκε ρητά ε, στην πρόταση και τη σύσταση περί κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 20 Δεκεμβρίου πέρυσι. Θα ήθελα τώρα να σας δώσω κάποια περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με τα ερωτήματα που θέσατε. Πρώτα απ' όλα, να επιζήσω την προσοχή σας, όπως ε, είπε η κυρία Ιντεβελτ, ε, στην πρόσφατη απόφαση της, ε, του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας, που, το οποίο επηρεάζει τη σημερινή συζήτηση. Το Ιρλανδικό Δικαστήριο ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ένα προδικαστικό ερώτημα σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Έντλμα Σύλληψη. Ένα Ευρωπαϊκό Έντλμα Σύλληψη που, προέρχεται από τι πολωνικές αρχές και αφορούν, αφορά ένα πολωνό υπήκο που συνελήφθη στην Ιρλανδία. Το Ιρλανδικό Δικαστήριο έθεσε το ερώτημα αυτό λόγω τη υπάρχουσας κατάσταση με το κράτος, του υποφέρου κράτου δικαίου στην Πολωνία και κατά πόσο ο άνθρωπος αυτός θα τύχει μια δίκαιη δίκη εφόσον επιστραφεί. Από εκεί και πέρα τώρα το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι αυτό που θα αξιολογήσει κατά πόσο η κατάσταση στην ε, Πολωνία μπορεί να επηρεάσει το Ευρωπαϊκό Σύλληψης. Δεύτερον, κυρία, η κυρία Ίντεβελ στο ερώτημά τη ε, ρώτησε πιο συγκεκριμένα πώς η παρούσα κατάσταση στην Πολωνία θα επηρεάσει τη λειτουργία των βάσεων δεδομένων. Το σύστημα ε, FIU-NET ε, με τις οικονομικές πληροφορίες, το ECRIS και το SIS. το SIS. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ε, δίκτυο για τα οικονομικά στοιχεία, το FIUNET, δεν είναι μια βάση δεδομένων της Europol. Είναι ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ε, μεταξύ των ε, υπηρεσιών οικονομικού εγκλήματος. Ακόμα και αν το διαχειρίζεται η Europol, πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο σύστημα, όπου οι πληροφορίες παραμένουν στα servers του FIU. Επίσης τα FIUs δεν διενεργούν έρευνες. Ο ρόλος τους είναι να κάνουν ανάλυση πληροφοριών για ύποπτες συναλλαγές που ε, λαμβάνουν από οικονομικές οντότητες και να διαδώσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης προς τις αρμόδιες αρχές εφόσον υπάρχει κάποια υποψία ξεπλήματος χρήματος ή χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών. Όπως ε, και τα περισσότερα FIU στην Πολωνία, ε, στην Ευρώπη ή το πολωνικό FIU δεν έχει ε, το καθεστώς επιβολής του νόμου. Είναι ένα διοικητικό, μια διοικητική δομή υπό το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ό,τι αφορά τώρα τη βάση δεδομένων έκρης. Η βάση δεδομένων έκρης είναι ηλεκτρονική, ένα ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για γρήγορη και αποτελεσματική ε, πληροφοριών σχετικά με τα ποινικά μητρώα ε, καταδικασμένων ε, υπηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2012 λειτουργεί το σύστημα αυτό. Ε, χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών, ποινικών διώξεων. Η Πολωνία είναι μεταξύ των κρατών μελών που είναι πλέον συνδεδεμένη με άλλα Σε σχέση με άλλα η Πολωνία λαμβάνει έναν μεγάλο όγκο ετοιμάτων για πληροφορίες σχετικά με τα ποινικά μητρώα ε, στα, εθνικά τους, στις ε, εθνικές μέσω του έκρης. Και η Πολωνία απαντάει στα αιτήματα αυτά με αξιόπιστο τρόπο και αυξάνεται ο αριθμός των μηνυμάτων που στέλνονται και λαμβάνονται από το έκρης σταθερά, σταθερή αύξηση από το 2012 έως το 2016. Σε ό,τι αφορά τώρα το σύστημα SIS, το σύστημα πληροφοριών Schengen, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζει να υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τα alerts τα οποία εκδίδει η Πολωνία. Και τέλος, ο αντίκτυπος για τη ε, ασφάλεια στην Ευρώπη εφόσον ένα κράτος μέλος αποτελεί αδύναμο κρίκο στα πλαίσια της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας. Όντως, σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να πει κανεί ε, ότι εφόσον στην αλυσίδα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας ένα κράτος μέλος αποτελεί αδύναμο κρίκο, αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Και θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι σε αυτό το πλαίσιο ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων είναι σημεία κλειδιά για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής, της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας. Η ασφάλεια και ο σεβασμός του κράτους, δικαίου και των θεμελιών δικαιωμάτων πάνε χέρι-χέρι. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεσμεύεται να προωθήσει τα κράτη, τα, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα διαφυλάξει. Ευχαριστώ πολύ όπως αντιλαμβάνομαι θα περιμένετε την απόφαση του δικαστηρίου στην περίπτωση αυτή. Ε, βεβαίως, περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου με μεγάλο ενδιαφέρον και θα αξιολογήσουμε την κατάσταση. Αλλά όλη αυτή την απόφαση περιμένουμε. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το τι κάνει η Κομισιόν αυτή τη στιγμή. Σόφι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Σύντομα, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επισημάνω στην κυρία Μορβάη πως μάλλον βρίσκεται σε λάθος σημείο της ημερήσια διάταξης. Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις εδώ και μόνοι μου να ήμουν εδώ πέρα, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Και το θέμα δεν αφορά την κυριαρχία της Πολωνίας, αφορά την, ε, τον νόμο και τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, την οποία έχουμε συνυπογράψει όλοι. Και η χώρα σας ήταν η πρώτη η οποία ακύρωσε την συνθήκη της Λισαβόνας. Πέρα από αυτό, ε, λυπάμαι τους καημένους ανθρώπους της Κομισιόν που στέλνουν εδώ πέρα για να κάνουν την ε, βρωμοδουλειά των επιτρόπων. Γιατί πρόκειται για ένα πολιτικό ζήτημα και έχω την αίσθηση ότι όταν ε, κάνουμε ερωτήσεις ε, προς την Κομισιόν και περιμένουμε απάντηση, είναι σαν να προσπαθεί κανείς να κολυμπήσει σε βούτυρο. Δεν, δεν πάμε πουθενά, δεν προχωράμε καθόλου. Δεν ήταν απάντηση αυτή στην Κομισιόν. Δεν ρώτησα για τρεις βάσεις δεδομένων και πώς λειτουργούν. Ρώτησα για το θέμα της αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα με την Κομισιόν, ε, όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα. Η Κομισιόν είναι κότα. Φοβάται να αγγίξει τα επίμαχα ζητήματα. Και περιμένει τώρα κάθε φορά το δικαστήριο να καθαρίσει το χάλι που έχει δημιουργηθεί. Και από την Κομισιόν και από το Κοινοβούλιο, για να είμαστε δίκαιοι. Έκανα την ερώτηση τον Οκτώβριο. Εν τω μεταξύ έβγαλε απόφαση ο Ιρλανδός δικαστής που ήταν απολύτως προβλέψιμη όπως, ήταν, όπως είναι προβλέψιμο ότι θα έχουμε και άλλα πολλά τέτοια προβλήματα. Ο Ιρλανδός δικαστής είναι μόνο η αρχή. Ε, πότε θα αναλάβει τις ευθύνες της Οικομισιόν. Το ανέφερε και η Μπάρμπαρα ΕΠΟ. Δεν είναι μόνο το θέμα εσείς έκουης και η βάση δεδομένων των οικονομικών αστυνομίων. Το θέμα είναι η δικαιοσύνη της Πολωνίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Συστήματος. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί επίσης ε, εφαρμόζουν και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εάν δεν θεωρείται λοιπόν πλήρως ανεξάρτητη η πολωνική δικαιοσύνη, κατά το οποίο μπορεί να συμπεράνουμε και για άλλα κρατημέλη κάποια στιγμή, τότε το σύστημα πάσχει. Και η Κομισιόν έχει ευθύνη για την τήρηση των συνθήκων. Θέλω λοιπόν μια πραγματική απάντηση. Όχι εγώ μόνο. Το θέμα αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλω μια πραγματική απάντηση και μετά θα επανέλθω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Έχουμε πέντε λεπτά μέχρι την ε, ψηφοφορία. Ε, προς τον κύριο Γιούρεκ Ζητήσατε τον λόγο μετά την συζήτηση. Α, κάτι άλλο. Ποιο? Α, υπάρχει και άλλο ένα θέμα. Με συγχωρείτε. Μετά την συζήτηση, μετά από αυτό το θέμα, είμαστε στο σημείο 7. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο θέμα είναι σχέδιο ψηφίσματος για το επαρκές επίπεδο προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα ιδιωτικότητας μετά από τα ευρήματα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έγγραφα που δημοσίευσε η Κομισιόν και η ομάδα εργασίας του άρθρου 29. Επίσης λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις μετά από την δημοσίευση αυτών των εγγράφων που θα επηρεάσουν την λειτουργία της ασπίδας αυτής και του επίπεδου προστασίας που πρέπει να διασφαλίζεται σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Παρουσιάζουμε εδώ πέρα λοιπόν τις συστάσεις προς την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και τις αρχές των ΙΠΑ έτσι ώστε η ασπίδα αυτή ιδιωτικότητα να εκπληρώνει τον στόχο της και να παρέχει το απαραίτητο επίπεδο προστασίας. Θα δώσω τώρα τον λόγο στους κοιόδησίτε. Και θέλει κάποιος άλλος. Α, όχι. Συγγνώμη. Ποιο είναι ο σκιώδης Α, Σόφη. Ωραία. πράγματα πέμπτη πρωί. Δεν θα πω πολλά πράγματα για το ψήφισμα, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχουν τόσοι λίγοι άνθρωποι εδώ ε, δεδομένου του ότι παράδειγμα τους κάνει μια εταιρεία όπως η Cambridge Analytica μεταφέρει δεδομένα είπα αυτό το καθεστώς στις είπα και όλο το σούσουρο που γίνεται για την εταιρεία αυτή και το facebook της μας θα περίμενα λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν είναι μυστικό πάντα θεωρούσα το ότι είναι ανεπαρκής αυτή η ασπίδα όπως και ο ασφαλής λιμένας το προηγούμενο σύστημα θα περιμένουμε και εδώ τι θα πει το δικαστήριο αλλά για να είμαστε συνεπείς ε, πρέπει να δούμε και τον σχεδιασμό αλλά και την εφαρμογή του συστήματο αυτού. Δηλαδή πόσα ψηφίσματα θα ευθύσουμε και θα λέμε ότι «Α, ναι, δεν τηρούνται όλοι οι όροι της συμφωνίας». Ε, πόσο θα περιμένουμε ακόμα για να γίνουν οι απαραίτητε ε, αλλαγές ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Το γεγονό ότι το χρησιμοποιεί η Cambridge Analytica και το Facebook και πολλές άλλες εταιρείε για παρόμοιους στόχους, νομίζω τα λέει όλα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ντάλτον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να υπογραμμίσω πόσο κρίσιμη σημασία είναι να δώσουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες, προστασία στου καταναλωτές και ασφάλεια στι επιχειρήσει στις επιχειρήσεις ό,τι αφορά προσωπικά δεδομένα. Μετά τον κανόνα, το κανόνα Safe Harbor δείχνει ε, ότι η ασπίδα που έχουμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα διεθνώς των πολιτών μας. Όταν κάποιος ταξιδεύει ε, εκτός των συνόρων θα πρέπει οι αξίες και τα δικαιώματα τα οποία εμείς περισπευόμαστε να διαφυλάσσονται. Τα δεδομένα λοιπόν αυτά προστατεύονται σωστά όπως λέει η έκθεση. Οι Αμερικανικές αρχές έχουν κάνει καλή πρόοδο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διαφόρων μηχανισμών, ε, την, ε, τις μηχανισμούς προσφυγών ε, και τις διαδικασίες εφαρμογής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως ξεκολουθεί να παρακολουθεί το θέμα του Privacy Shield έτσι ώστε οι πάνω από 2.000 εταιρείε ε, ε, να έχουν κατάλληλη προστασία. Υπάρχει ένα σύστημα στι ΗΠΑ το οποίο θεσπίζεται, αλλά πρέπει εμεί να υποπτεύουμε. Υπάρχουν μια σειρά από συστάσεις τι οποίε θα ήθελα λοιπόν να συμπεριληφθούν σε αυτή την έκθεση. Στο εμπορικό επίπεδο, το, το Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου θα πρέπει ε, ε, να, μην, να μην αφήνει τι εταιρείε να δημοσιοποιούν ότι έχουν λάβει το πιστοποιητικό του Privacy Shield πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρέπει να υπάρχουν λεπτέ γραμμέ, ε, παραδείγματο χάρη ε, για τα δεδομένα ε, HR. Ε, θα χρειαστούμε πολιτική βούληση για να υπάρξει εμπιστοσύνη και αποτελεσματική διοικητική του Privacy Shield, ε, αποτελεσματική εφαρμογή. Θα πρέπει επίση να υπάρχει και ένα ombudsman, ένα διαμεσολαβητή σε ό,τι αφορά το Privacy Shield που θα έχει συγκεκριμένε αρμοδιότητε ε, και θα ασχολείται ε, γενικότερα με τα ζητήματα ε, ελευθεριών. Χρειαζόμαστε επίση υψηλά ποιότητα βάσει δεδομένων, των δεδομένων, προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αλλά αυτό θα επηρεάσει και την ανταγωνιστικότητα της Ένωση. Θα συνεργαστούμε με τους ε, και είμαι σίγουρο ότι θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό ψήφισμα. Η ε, κυρία Γκιουλιάν έχει το λόγο. Ναι, θα μιλήσω στα αγγλικά στη συνέχεια στο όνομα της Μπρίγκη Τζίπελ που μόλις μου έστειλε ένα μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον Πρόεδρο για αυτό το σχέδιο κειμένου. Είναι πολύ στροπημένο κείμενο το οποίο ε, δεν παραβλέπει μια σειρά από ανησυχίες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά το Privacy Shield. Εδώ περιλαμβάνεται πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι δεν λειτουργεί απολύτως το Συμβούλιο Παρακολούθησης, δεν έχουν ακόμα οριστεί όλα τα μέλη. Δεύτερον, η, Ευρωπαϊκή, η Αμερικανική κυβέρνηση ε, δεν έχει ακόμα ορίσει έναν διαμεσολαβητή, παρότι αυτό είναι προαπαιτούμενο του κοινωνικού δικαίου. Επίσης, οι πρόσφατες ε, αποκαλύψεις ότι το Facebook και η Cambridge Analytica έχουν ε, λάβει το πιστοποιητικό του πράγμα Shield αλλά έχουν κάνει κακή χρήση δεδομένων και έχουν ευνοήσει και επηρεάσει πολιτικές καμπάνιες ε, αυτά πρέπει να, να ληφθούν υπόψη πάντως κατά τα άλλα η πρόταση είναι καλή τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βος Ευχαριστώ Ευχαριστώ που μου δώσετε και τον λόγο πρόταση που κάνουμε εδώ είναι κάπως ε, πολύ αρνητική. Με το Safe Harbor και το πέρασμα στο Privacy Shield δημιουργήσαμε κάτι που πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση και είδαμε ότι τελικά πρώτον είχαμε αρκετή πρόοδο και δεύτερον ε, κάποιες θετικές εξελίξεις. Το ότι τώρα προέκυψε το Facebook και το Cambridge Analytica είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ να αλλάξει αυτό το οποίο κάνουμε. Δηλαδή είναι, δεν εμποδίζουμε καμία εγκληματικότητα με τους ε, νόμους. Ε, πρέπει όμως ε, να την αντιμετωπίζουμε και το ερώτημα είναι τελικά τι μπορούμε να βελτιώσουμε στην πλευρά του ελέγχου. Θεωρώ λοιπόν ότι το Facebook και η όλη αυτή η κατάσταση έδειξε πως ε, κάτι κάνουν και στις ε, είπα δεν ότι κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Και ακριβώς εμείς επειδή έχουμε την, τον κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων και το Privacy Shield είμαστε πολύ πιο εστιασμένοι. Οπότε, η αξιολόγηση του Privacy Shield ε, καθ' αυτού νομίζω ότι είναι θετική. Οπωσδήποτε δεν είναι ωραίο το ότι δεν έχουν στελεχωθεί διάφορες επιτροπές ε, Εντάξει, υπάρχει κάποιος ο οποίος ε, τα κάνει αυτά προσωρινά, δεν υπάρχει κενό λοιπόν Εντάξει, καλό είναι να οριστικοποιηθούν βεβαίως τα πράγματα. Αλλά βεβαίως, εντάξει, δεν υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες. Πρέπει όμως να υπάρξουν αυτοί οι διορισμοί και να δούμε το ότι θα πρέπει και η Αμερικανική κυβέρνηση να παίρνει στα σοβαρά τα όσα έχουμε συμφωνήσει. Αλλά νομίζω ότι το Privacy Shield είναι ένα καλό παράδειγμα για το ότι μπορούμε να πάμε σε μια λογική κατεύθυνση. Εντάξει, ίσως όχι 100% από την αρχή. Αλλά θα έχουμε κάθε χρόνο και την σχετική έκθεση και μπορούμε να βελτιώνουμε τα πράγματα λίγο λίγο. Μην είμαστε λοιπόν υπερβολικά αρνητικοί γιατί έχουμε την εντύπωση αυτή ε, από το facebook ότι δεν λειτουργούν τα πράγματα αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι σημάδι ακριβώς του ότι όντως λειτουργούν. Η κατάχρηση τώρα βεβαίως δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί. Ε, πρέπει να είμαστε κάπως πιο θετικοί για να είμαστε περήφανοι για αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ένστ. Ε, ίσως εμείς οι αριστεροί να είμαστε κάπως πιο απεσιόδοξοι. Ε, έχουμε διαβάσει όλη την ίδια έκθεση. Γιατί δεν ξέρω. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μπορεί να διαβάσαμε άλλο εγγραφό. Εγώ βλέπω εδώ σοβαρή κριτική από την Επιτροπή του άρθρου 29. Λέει σοβαρές ανησυχίες μιλάει για επανεκκίνηση των συζητήσεων που χρειάζεται, χρειάζεται σχέδιο δράσης, ο διαμεσολαβητής ε, είναι και η συμπλήρωση όλων αυτών. Και είναι σαφές ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η ασπίδα προστασίας δεν είναι ασπίδα προστασίας. Είναι φιλοσικής. Αυτό βλέπουμε και όπως και να το πούμε, μπορούμε να το πούμε πιο Ωραία, εντάξει δεν άγγε να έχουμε μυρολατρεία, αλλά ξεκαθαρά εδώ πέρα είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν λυθεί, δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Και ο ανεξάρτητος δημοσιολογητής, όπως λέμε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία δικλείδα ασφαλείας. Ε, όταν δεν έχει γίνει καμία αλλαγή, με τι να είμαστε ικανοποιημένοι. Υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου, κάτι θυμάμαι για το Safe Harbor. Και είπαμε τότε ότι πρέπει να το αλλάξουμε και λέει η Κομισιόν ναι θα το κάνουμε και καταλήξαμε με αυτό το... με αυτή την ασπίδα προστασίας. Έτσι, χοντρικά έτσι γίναν τα πράγματα. Α, τελικά δεν έγιναν και πολλά πράγματα. Θέλω να ακούσω την Κομισιόν τι θα κάνει με βάση αυτή την παρουσίαση που δεν είναι και θετική, έτσι. Τι θα γίνει με το σχέδιο δράσης. Τι σκοπεύει να συζητήσει. Η κυρία Κιούροβα μας υποσχέθηκε κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν θα μας κοροϊδεύουν. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μας ε, κοροϊδεύουν. Αν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες μας θέση, δεν θα ήταν τόσο χαλαρές. Το Facebook αποδεικνύει και ελπίζω και ο Σάγκερμπερκ να έρθει και εδώ πέρα Δείχνει λοιπόν η υπόθεση το πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και ποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Και δεν ε, λύνεται τίποτα. Γι' αυτό θέλω να ακούσω από την Κομισιόν τι σκοπεύει να κάνει. Λοιπόν, Ευχαριστώ να ζητήσω από τους υπόλοιπους βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Μητροπή Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να λάβουμε το λόγο. Κάποια σχόλια. Καταρχάς, νομίζω συμφωνούμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αυτό λέει και η έκθεσή μας μετά την αιτήσια αποτίμηση της ασπίδας προστασίας, της ιδιωτικότητας. Όταν εγκρίθηκε βέβαια η απόφαση, αποφασίσαμε να υπάρχει ένα τάδε επίπεδο προστασίας. Ελέγξαμε κατά πόσο ισχύει, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αυτό ε, το είδαμε και στην συνέχεια των εξελίξεων μετά την δημοσίευση της ετήσιας αποτίμηση και σε σχέση με κάποια ζητήματα που εντόπιζε η έκθεση. Υπάρχει μάλιστα και συνέπεια απόψεων με κάποιες από τις ε, αρχές παρακολούθησης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων με τις οποίες συνεργαζόμαστε κιόλας για την εκπόνηση της εκθεσής μας. Όπως είπα όμως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και για τον ε, ε, εκκρεμή διορισμό του μόνιμου διαμεσολαβητή διαμεσολαβήτριας ε, παρόλο που υπάρχει κάποιος που ασκεί καθήκοντα διαμεσολαβητή προσωρινά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει. Περιμένουμε όμως εδώ και ένα χρόνο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ με τις συνομιλίες της και τις επαφές της με τις Αμερικανικές Αρχές και με συναντήσεις όπως τον τελευταία το Μάρτιο λόγω χάρη, τονίζει αυτό ότι χρειάζεται να διοριστεί δημοσιολαβητής Είναι σημαντικό να γίνει ο διορισμός αυτός, διότι αλλιώς θα έχουμε νομικό πρόβλημα. Και θα είναι και σημαντικό ε, δείγμα ότι αποδίδουμε τη δέουσα προσοχή στο θέμα αυτό για να υπάρξει και ένα κλίμα εμπιστοσύνη. Θα πρέπει οι αρχέ να δείξουν ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ασπίδα προστασία του ιδιωτικού βίου. Ε, άλλοι διορισμοί επίση έγιναν όπως το Εποπτικό Συμβούλιο, το πλέον για την ε, ιδιωτικότητα. Το τι κλαμπ θα πρέπει να φτάσει ακόμη σε πλήρη απαρτία βέβαια, δηλαδή να γίνει πλήρης ε, σύνθεση, ε, αν και έχουν ήδη διοριστεί τρία μέλη. Έχουν γίνει ακροάσεις τους, οι συνεντεύξεις τους και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουν ε, και θα διοριστούν και οι υπόλοιποι δύο. Δεν έχει λοιπόν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του Συμβουλίου, το εξηγούμε όμως και στην ετήσια έκθεση. Δεν είναι ότι δυσλειτουργεί αυτή τη στιγμή το P-Club, αλλά συναντήσαμε εκπροσώπους του και μας είπε ότι προχωρεί η δουλειά τους και σε σχέση με το αμερικανικό σύστημα και το σχετικό νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πάντως ελπίζουμε οι διορισμοί ότι θα γίνουν γρήγορα. Συμφωνώ και με αυτό που ο κύριος Ντάλτον πρέπει η αρχή που είναι υπεύθυνη για την ε, εφαρμογή του, της ασπίδας προστασίας και το τμήμα που είναι η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία να αναλάβουν περισσότερη δράση. Αυτά ε, τα είδαμε και στην υπόθεση του Facebook και της Cambridge Analytica. Και σίγουρα μας απασχολεί το κατά να χρησιμοποιούνται σωστά τα προσωπικά δεδομένα, όπως και άλλους. Αλλά θα πρέπει ε, να είναι σε επιφυλακή όσοι ασχολούνται με τα εμπορικά θέματα. και να κάνουν τον σχετικό έλεγχο εγκαίρως. Όπως επίσης και η Αμερικανική Επιτροπή που παρακολουθεί το θέμα αυτό έχει κάνει τις σχετικές έρευνες, είχε ερευνήσει για το Facebook Υπήρξε κάποιο διακανονισμό τότε και αυτή τη στιγμή ελέγχει κατά πόσον ο διακανονισμό εκείνο παραβιάστηκε πάλι. Η αίσθηση λοιπόν κάνει τη δουλειά τη, αλλά δεν θα πρέπει να ασχοληθεί μόνο με το Facebook, επειδή αυτό απλώ πήραμε χαμπάρι, αλλά να κοιτάξει με την ίδια προσοχή και άλλες εταιρείε που οι πρακτικέ του μπορεί να είναι αθέμητες. Ιδίω εκεί που υπάρχει περίπτωση υπεξαίρεση και κακής ε, χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την ετήσια έκθεσή της. Δεν ε, χρειάστηκαν μόνο συναντήσεις δύο ημερών, ας πούμε. Έγιναν επανειλημμένο συναντήσεις εκπροσώπων από διάφορες ε, αμερικανικές αρχές και αμερικανικούς φορείς, με τους δικούς μας. Ετοιμάσαμε ερωτηματολόγια και ούτω καθεξής και εκτοτέ ε, αφότου εκδώσαμε τις συστάσεις μας και πάλι υπήρξαμε πολύ δραστήριοι και σε επίτροπο επιτρόπων αλλά και σε τεχνικό. Είχαμε πολλές συναντήσεις μαζί τους. Ναι, πρόεδρος. Εντάξει. Σας παρακαλώ όμως, ολοκληρώστε. Ναι. Ε, μας είπαν ότι θα ληφθούν κάποια μέτρα για να αντιμετωπίσουν ε, αυτά που τους θέσαμε ως προβληματισμούς, ιδίως για τις εμπορικές πτυχές και σε στενή συνεργασία με τις αρχές προστασίας δεδομένων. Είναι και αυτό σημαντικό. Και το καλλιεργούμε ώστε να καταλήξουμε σε μια κοινή πορεία και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μα. Για να βεβαιωθούμε ότι υποθέσει όπω αυτέ του Facebook με την Cambridge Analytica θα, θα ξανασυμβούν. Uh, τώρα η Σοφή Ιντεφελτ για να συνοψίσει. Ε, ναι, αυτό μπορώ να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κοντά στο μηδέν σε ό,τι αφορά τις, δυνατότητε δυνατότητες Ε, έχουμε την ίδια συζήτηση που είχαμε και για την ασφαλή λιμένα, το Safe Harbor. Δεν έμαθαν δεν έμαθαν να ακούν τους εμπειρογνώμονες, τους ειδικού. Δεν έχουμε τόσα παραδείγματα πλέον όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αγνόησε ε, τις απόψεις του EDPS, ε, άλλων ε, ειδικών και τελικά αυτά τα ζητήματα αναπόφευκτα πάνω στο δικαστήριο και εκεί χάνουμε. Πόσες φορές μπορεί να κάνει κανείς το ίδιο λάθος. Είναι ενδιαφέρον το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος αναφέρθηκε στην Cambridge Analytica και στο Facebook, διότι και εγώ τα ανέφερα ως παράδειγμα για να αποδείξω πως το Privacy Shield δεν λειτουργεί. Ο πρόεδρος Τραμπ εποφελήθηκε από το γεγονός ότι δεν λειτουργεί προφανώς. Μια και το Cambridge Analytica και το Help Facebook τον βοήθησαν να κερδίσει τι εκλογέ. Τι, νόη, τι, τι ενδιαφέρον έχει λοιπόν ε, ο ίδιος για να λειτουργήσει. Εγώ μπορεί να είμαι λίγο ντεμοντέ, αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχει μια συμφωνία, ένας νόμος, δεν ζητούμε ευγενικά από την άλλη πλευρά ε, να εξετάσει το κατά πόσο θα, σε, σεβαστεί τη συμφωνία. λέμε ότι είτε σέβεται τη συμφωνία είτε ε, δεν υπάρχει συμφωνία. Ίσως να είναι λίγο ξεπερασμένη η λογική αυτή. Ε, μα λοιπόν, συστάσεις, αιτήσεις Όχι. Όχι, ή θα δεχτούν τη συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει privacy shield. Ε, και εδώ η Κομισιόν έχει καθήκον να παίρνει στους Ευρωπαίους πολίτες, όχι προς την Αμερικανική κυβέρνηση, προς τους Ευρωπαίους πολίτες, να υπερασπιστεί τα δικαιώματά τους. Και αποτύχαμε ικτρά με την Cambridge Analytica και με το Facebook και μάλλον και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που καλύπτει από το privacy shield. Λοιπόν, ε, πρέπει να εξηγήσετε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που έχετε εξηγήσει ως τώρα. Uh, Ευχαριστώ. Να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 23 Απριλίου του 2018. Θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία σε τρία λεπτά.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

I, I,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

Λοιπόν, ελπίζω να έχετε τις κάρτες για να ψηφίσετε. Θα αρχίσουμε με το σχέδιο γνωμοδότησης ε, για το scoreboard ε, την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη τον πίνακα δηλαδή η Σίλβια Κιγιάμ είναι η συγγήτρια Γιώμη είναι η συγγήτρια συγγνώμη δεν θέλετε το λόγο δεν θέλετε λόγο κυρία Κιγιώμη Λοιπόν, συμβασμός 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. 15. Άχι η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεκαεπτά. Άχι η ψηφοφορία. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Συμβασμός 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 4. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 10. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 3. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 44. Συγγνώμη, συμβιβασμός 5. Συμβιβασμός 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ. Ε, άρχισε η ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας ψηφοφορία ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία απορρίπτεται. Συμβασμός 7. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, παραπομπή 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Εκτιμώντα τώρα. Ή ε, μάλλον, συμβασμό 12. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Monica too late. We finished voting. Ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στη μέση διάταξη είναι μια ενημέρωση στην Επιτροπή για την πρόταση κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση των διαταγών κατάσχεσης και ε, παγώματος. Ε, παρακαλώ, ησυχία. Κατάσχευση και δίμευση, συγγνώμη. Ε, ξεκινάμε την εκτέλεση του επόμενου σημείου ψηφίστηκε στην Επιτροπή Ελευθεριών ε, τον Ιανουάριο του 2018. Είχαμε τον Τρίλογο. Οι βασικές αλλαγές, οι διαφορές μεταξύ των συνομοθετών ε, ε, σημειώθηκαν σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες, τους λόγους μια αναγνώρισης, την κοινωνική επαναχρήση των ε, δημιουργημένων περιουσιακών στοιχείων, τα νομικά μέσα, η δικλείες ασφαλείας, καθώς και εφαρμογή ε, σχετικά με την, την σχετικά, καθώς και η ημερομηνία εφαρμογή του κανονισμού. Έχετε το λόγο, κυρία εισηγήτρια, κυρία Γκρίσπεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως προηγουμένως θα προσπαθήσω και εγώ να, να ανοίξω την πόρτα γιατί δεν το μικρόφωνο. Α, τέλος πάντων να σας ενημερώσω για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων στους τριμμένους διαλόγους για το θέμα αυτό. Θυμήσατε μόλις τον τίτλο «Ευρωπαϊκός κανονισμός για την αμοιβαία αναγνώριση των διαταγών παγώματος και δίμευσης ε, περιουσιακών στοιχείων που είναι προϊόν εγκληματικών ενεργειών. Ε, θέλουμε συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, ώστε να μπορούμε να δημεύουμε ή να κάνουμε κατάσχεση και πάγωμα πολύ γρήγορα και αποτελεσματικό κυρίω των προϊόντων οικονομικού κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από μνήμης να σας πω ότι πάνω από 98% ε, των κερδών του παράνομου εγκλήματος αυτή τη στιγμή δεν δημιουργούνται ούτε κατάσχονται αλλά μένουν στα χέρια των, εγκληματών, των εγκληματιών. Ε, από τεχνικής λοιπόν πλευράς το εργαλείο αυτό είναι εντελώς ε, απαραίτητο και το καλωσορίζουμε. Μερικές υπενθυμίσεις για το χρονοδιάγραμμα, τα γενικά σχόλια και την πρόοδο των εργασιών μας δηλαδή τι συζητιέται στο πλαίσιο του τριμέρους διαλόγου. Χρονοδιάγραμμα. Ψηφίσαμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ με βία πλειοψηφία το θέμα αυτό τον Ιανουάριο του 2018. Πολύ γρήγορα ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει σε τριμερή διάλογο μετά, στις 23 Ιανουαρίου ο πρώτος. Μετά είχαμε δύο τριμερείς, δύο τριμερείς πολιτικούς διαλόγους και τέσσερις τεχνικούς. Και την επόμενη εβδομάδα ξανά έχουμε τριμερή διάλογο στο Στρασβούργο. Μερικά γενικά σχόλια για τη γενική προσέγγιση. Οι διαπραγματεύσει οδεύουν καλώ, με καλό πνεύμα συνεργασία και εδώ να υποφεληθώ διότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία με του συναδέλφου Κιώδη, οι οποίοι με βοηθούν για τη σύνταξη του θέματο αυτού, της έκθεσης αυτής. Ε, η Βουλγαρική Προεδρία έχει την πρόθεση να ολοκληρώσει εφόσον ε, γίνεται την εξέταση του θέματος στο εξαμεινό τη, άρα επιδεικνύει και εκεί την απαραίτητη και εκείνη την απαραίτητη προθυμία και την ευχαριστώ και αυτήν και πολύ γρήγορα να πω ότι για τα τρία θεσμικά όργανα έγινε σαφές δεν συμβαίνει πάντοτε είναι κάτι το θετικό. Να θέλουμε ένα εργαλείο σαφές, συνεπές, πρακτικό και εύκολο να λειτουργήσει. Δεν είναι πάντοτε αυτό που συμβαίνει σε τέτοιες ε, πρωτοβουλίες. Ως προς την ε, μορφή του κειμένου. Θέλαμε να είναι κανονισμός ε, το κείμενο και όχι οδηγία. Στην αρχή τα πράγματα ήταν λίγο χάος. Έπρεπε να συζητήσουμε και να πιέσουμε για να μπορέσουμε όλοι να ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή. Το κοινοβούλιο ήταν συσπηρωμένο, οπότε ευτυχώς αυτό ήταν ένα επιχείρημα για να πείσουμε για τους υπολείπους. Τι καταφέραμε να γίνει τελικά αυτό που θέλαμε. Ως προς τη διαδικασία. Βεβαίως το Κοινοβούλιο ε, επαγρυπνεί ώστε οι δικονομικές εγγυήσεις να ληφθούν σοβαρά υπόψη και κάτι που συζητάτε πολύ αλλά δεν είχαμε χρόνο να το αναπτύξουμε και δεν καταλήξαμε και σε συνένεση μεταξύ μας ε, για το τι θα ήθελε το Κοινοβούλιο είναι το θέμα της συμπερίληψης μιας ρήτρας μη αναγνώρισης, μη εκτέλεσης δηλαδή των αποφάσεων για πάγωμα ή δίμευση όταν αυτές βασίζονται σε ε, μη ε, σεβασμό, απουσία σεβασμού των ε, δικαιωμάτων. Είναι νομίζω λογικό, είναι μια απέτηση πάγια και θεμητή θεωρώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έχουμε εκφράσει εδώ και χρόνια, οπότε Μπορεί να δυσκολευτούμε λιγάκι στις διαπραγματεύσεις, όμως θα φροντίσουμε να ε, παραμείνουμε οκίνητοι. Επίσης, ε, σε κάτι άλλο που συμφωνούμε όλοι οι σκιώδες μεταξύ μας, ε, είναι ότι η διαδικασία θα πρέπει να είναι ταχεία. Είναι ένα άλλο σημείο επί του οποίου θα πρέπει να συζητήσουμε και άλλο με το Συμβούλιο διότι το Κοινοβούλιο έχει προσθέσει τέτοιες ε, προθεσμίες ώστε να υπάρχει και ταχύτητα και ε, διαφάνεια και συνοχή στη χρήση του εργαλείου. Εδώ πρέπει να γίνει μια περισσότερη προσπάθεια και από την το πλευρά του Συμβουλίου που δεν ήταν τόσο σαφές. Το επιδιώκουμε λοιπόν σε συνεργασία με τη Βουλγαρική Προεδρία. Και τέλος τρίτο η τέταρτο στοιχείο, και θα ολοκληρώσω με αυτά, είναι ότι θέλουμε να υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο κοινωνική, η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των ε, δημευμένων, υπαγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Εδώ αναζητούμε μια κοινή θέση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, διότι το Συμβούλιο ε, έχει δώσει μια ε, περίοπτη θέση ε, στην όλη στρατηγική, στην αποζημίωση προς τα θύματα ε, και την ε, αποζημίωση των ενώσεων θυμάτων, θυμάτων τέτοιων περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος. Έτσι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, οι διαπραγματεύσει μέχρι τον επόμενο γύρο τριμερού διαλόγου την ερχόμενη εβδομάδα. Βεβαίω και πάλι να ευχαριστήσω του συναδέλφου και είμαι στη διάθεσή του για να συνεχίσουμε τι κοινέ μα προσπάθειε. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ε, κυρία Σπινέλη θέλει το λόγο. Συνάδελφοι, εάν θέλετε το λόγο, παρακαλώ να σηκώνετε το χέρι σας, ε, αλλιώς δεν σας βλέπω και θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ναι. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ από καρδιά στην ε, κυρία Γκρισπέκ για όσα έχει κάνει. Θέλω απλώς να παρατηρήσω το εξή. Ο κανονισμός αυτός είναι άκρος σημαντικός και το ξέρει πολύ καλά η Ναταλή, ειδικά για τη χώρα μου, όπου υπάρχει πραγματικά ζήτημα και ανάγκη δίμευσης και κατάσχεσης ε, περιουσιακών στοιχείων που έχουν στα χέρια τους οι πολλές μαφίες της χώρας. Ε, μαφίες που σε κάποιες περιοχές και περιφέρειες της Ιταλίας κάνουν κανονικά κουμάντο. Ε, να τονίσω ότι αυτό που συνέβη στη Σλοβακία με τη δηλοφωνία του Γιάνν Κούτσιακ που μάλλον δολοφονήθηκε από καλαβρέζικο πλοκάμι της ε, τοπικής μαφίας. Αυτό αποδεικνύει ότι ο κανονισμός πρέπει να είναι ευρωπαϊκός. Θέλουμε τέτοιο κανονισμό, διότι το οργανωμένο έγκλημα και η μαφία είναι πολύ καλά διοργανωμένοι σε διακρατικό επίπεδο. Ευχαριστούμε λοιπόν Ναταλή για τη δουλειά σου και θα είμαστε ε, δίπλα σου για να προτείνουμε ε, χρήσιμες ιδέες. Ωραία, συνάδελφοι. Τελειώνει αυτή η συζήτηση. Επόμενο τριμερής διάλογος στις 18 Απριλίου 2018. Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας ε, στις ε, Βρυξέλλες 25 Απριλίου. 9 με 12,5 και 2,5 με 6,5 και στις 26 Απριλίου. 9 με 12,5 και 2 με 5,5 το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.